Monsieur, Monsieur Razi, bienvenue. Καλώς ήρθατε κύριε Ράζη. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε την ικανοποίηση να υποδεχθούμε σήμερα το απόγευμα τον κύριο Ράζη, του υποψήφιο τελεξιστικού διευθυντή για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Χαιρετίζω και τους καθηγητές Λεμέρ και που παρευρίσκονται εδώ σήμερα να σας υπενθυμίσω τη μορφή της ακρόσης μας. Θα δώσω καταρχήν το λόγο στην κύριο Ράζη για 10 λεπτά για να μας παρουσιάσει το σχέδιό του, να μας πει όσα θέλει να μας καταθέσει εδώ. Κατόπιν θα ακολουθήσουμε την διαδικασία ping-pong, δηλαδή ένα λεπτό για την αρχική ερώτηση, δύο λεπτά για την απάντηση του κυρίου Ράζη, 45 δευτερόλεπτα για συμπλήρωμα στην αρχική ερώτηση και πάλι ένα λεπτό για τον κύριο Ράζη για να απαντήσει. Αυτή η ανταλλαγή θα γίνει σε τρία στάδια. Ένα πρώτο στάδιο με τα ερωτήσεις από τους συντονιστές, δεύτερο στάδιο με οκτώ ερωτήσεις και τρίτος γύρος με έξι ερωτήσεις που θα μας οδηγήσουν σε ταχύτερη διαδικασία. Θα έχουμε πιο γρήγορε, πιο σύντομε ερωτήσει εκεί. Αυτή η ακρόση του κυρίου Ράζη γίνεται στο πλαίσιο της γνωμοδότησης που μπορεί να η Επιτροπή μας για την υποψηφιότητά του. Κατόπιν τη γνωμοδότησής μα, η διάσκεψη των Προέδρων θα λάβει μια επίσημη θέση, η οποία θα διαβιβαστεί στο Συμβούλιο, στο Διοικητικό Συμβούλιο της EMA, ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, που θα πρέπει να διορίσει τον εκτελεστικό διευθυντή. Έτσι λοιπόν, ελπίζω όλα να είναι σαφή. Σας δίνω το λόγο κύριε Ρέζη για 10 λεπτά. Thank you. Ε, Mr. Chair, honorable... Ε, Πρόεδρε, Αξιότιμα μέλη, είναι μεγάλη τιμή που βρίσκουμε σήμερα εδώ ενώπιον ε, της Επιτροπής σας. Είναι μία εμπειρία την οποία δεν θα μπορούσα να είχα καν ονειρευθεί πριν από μερικού μήνες. Και είμαι πολύ ευτυχής που μου δίνεται η ευκαιρία να ε, σας ε, συστηθώ εκτός από τις προκλήσεις που ενδεχομένως θα συναντήσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων οπότε θα δοθεί ευκαιρία να ξανασυναντηθούμε ε, ελπίζω να εκδοθούν και άλλες ευκαιρίες συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από το οποίο αναμένω ενθάρρυνση, ιδέες, προτάσεις και συμβουλές. Θα ήθελα να μιλήσω σήμερα στη μητρική μου γλώσσα, ίσως για μία από τις τελευταίες φορές, διότι εάν αναλάβω το έργο αυτό του εκτελεστικού διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, θα μπορέσω ως ε, υπάλληλος των Ευρωπαϊκών, ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μιλάω μόνο σε επίσημες γλώσσες. Έτσι λοιπόν, όπως ε, σας είπα, για τα επόμενα χρόνια εγώ βλέπω κάποιες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε διάφορα επίπεδα. Φυσικά θα υπάρχουν και περικοπές στον προϋπολογισμό και θα υπάρχει διεύρυνση της εντολής, θα, υπάρχει, θα προβλέπεται αύξηση του αυθούς εργασίας, ε, βραχυπρόθεσμα βάσει της νέας νομοθεσίας για τη φαρμακοπεραγρύπνηση και για ε, τα ψευδεπίγραφα φάρμακα. Ε, δημιουργηθεί και η νέα επιτροπή για τη φαρμακοπεραγρύπνηση. Έτσι λοιπόν θα έχουμε 7 επιτροπές στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και σίγουρα ε, θα προσθέσουν πολυπλοκότητα στη λειτουργία του οργανισμού και θεωρώ ότι τρόπος ε, λειτουργίας ε, των διάφορων επιτροπών θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να αποσαφινιστεί. Αυτές ε, είναι προκλήσεις ε, διαχείρισης, ε, business as usual και καθημερινά κάθε αρμόδιος κάποιας εθνικής υπηρεσίας αντιμετωπίζει τέτοια φαινόμενα καθημερινά και σε διαφορετική κλίμακα. Όμως υπάρχει και ένα ανώτερο επίπεδο προκλήσεων που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. το χάρη η Ευρώπη χάνει σε ανταγωνιστικότητα ενότητα εναντί των αναδυόμενων χωρών από τις χώρες BRIC, Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα. Και σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις ε, στις κλινικές έρευνες ε, και αυτό θέτει πρόβλημα εναρμόνισης ε, της ρύθμισης των κλινικών δοκιμών μέσω των διάφορων κρατών μελών. Είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε επίσης ότι η κλινική έρευνα δεν αντιμετωπίζει μόνο το πρόβλημα της επένδυσης Αν εμείς... Ε, σκεφτούμε την έλευση των φαρμακών της επόμενης γενιάς, τα ένα φάρμακα, όπως το αποκαλούμε, τον οποίο οι θεραπευτικοί στόχοι θα καθορίζονται όλο και περισσότερο βάση σε φαρμακογενετικά κριτήρια, τότε καθίσταται προφανές ότι τα φάρμακα αυτά θα μελετώνται βάσει ενός πληθυσμού που πράγματι θα λαμβάνει αυτό το φάρμακο. Έτσι λοιπόν δεν θα μπορούμε να θεωρούμε ότι είναι καλό ότι μας έρχεται από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και φυσικά υπάρχουν και τα ηθικά προβλήματα. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι το θέμα της ε, απόκλησης ε, κρίσεων ε, που γίνεται μέσω της, μεταξύ της αξιολόγησης κινδύνου και ωφέλους που γίνεται από τον ΕΟΦ και της συγκριτικής αποτελεσματικότητας που θα χρειαστεί να υποστηρίξουν στη συνέχεια διάφοροι οργανισμοί και κατόπιν θα έχουμε και την λεγόμενη αξιολόγηση της τεχνολογίας της υγείας. Εδώ υπάρχουν όλο ένα και περισσότερες επικλήσεις και φυσικά προκύπτει εμπόδιο στις, ε, ε στην καινοτομία ε, και στις επενδύσεις και τελικά στην πρόσβαση των ασθενών ε, στα φάρμακα. Ο κατάλογος θα μπορούσε να είναι πολύ πιο μακρύς. Ένα παράδειγμα θα μπορούσε να είναι η ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά, η διαθεσιμότητα των κτηνιατρικών φαρμάκων, ε, η διαχείριση ε, της αξιολόγησης ε, της παραδοσιακής ιατρικής, τα σύνορα αυτά γίνονται όλο ένα και πιο δύσκολο να τα διαχειριστούμε, αλλά δεν θέλω να σας αναφέρω τώρα όλο αυτό το κατάλογο. Βέβαια, ε, ο ΕΟΦ συνεργάζεται στενά με την Κομισιόν και το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν θα πρέπει να μπορούν να βασίζονται στην εύρωστη ε, επιστημονική γνωμοδότηση του ΕΟΦ ε, σε ό,τι αφορά τη δημόσια υγεία. Γι' αυτό το θέμα, ε, λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε πολύ μεγάλη διαφάνεια και πάντοτε να διαχειριζόμαστε ορθά τα σύγκρουση συμφερόντων. Η πραγματική πρόσκληση είναι να προβλεψούμε τις μελλοντικέ εξελίξεις γιατί θα προκύψουν. Ε, Παραδείγματο χάρη, εξέλιξη στην επιστήμη θα μπορούσε να μα οδηγήσει στο να ρυθμίσουμε φάρμακα που να βασίζονται σε εντελώ καινούργια συστήματα χορήγηση των φαρμάκων. Παραδείγματο χάρη, έχουμε και την ενοτεχνολογία. Και να προβλέψουμε την χρήση βιοδικτών και την αξιολόγησή του. Θα μπορούσαμε έτσι επίση να βρεθούμε ε, στο να χρειαστεί να αξιολογήσουμε θεραπείε με φάρμακα που χορηγούνται με νέε τεχνικέ. Έτσι λοιπόν η σημερινή διαδικασία που αξιολογεί τον κινδύνο ενό και μόνου φαρμάκου θα μπορούσε να είναι εντελώ απαράδεκτη, να μην εφαρμόζεται καθόλου. Έτσι λοιπόν ο ΕΟΦ θα έπρεπε να είναι σε θέση να χειριστεί αυτό το μέλλον με του κανόνε που θα καθορίσουν Κομισιόν και Κοινοβούλιο. Με άλλα λόγια, εγώ πιστεύω ότι οι κανόνε τη δεύτερη χιλιετίας θα μπορούσαν να μην εφαρμόζονται πλέον στα φάρμακα που θα αναπτυχθούν στην τρίτη χιλιετία. Αλλά πριν ε, ακόμη να περάσουμε στη διαχείριση του μέλλοντο, νομίζω ότι πρέπει να καλύψουμε τα παλιά κενά. Η ανάπτυξη των φαρμάκων, ο σχεδιασμό θα πρέπει να ε, να καλύπτει περισσότερο, να φροντίζει περισσότερο να καλύψει τις απαιτήσεις ορισμένων πληθυσμών όπως των παιδιών ή των ηλικιωμένων και θα πρέπει επίσης να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ε, στις κλινικές μελέτες. Συμπρασματικά εγώ πιστεύω ότι αν η ΕΜΕΗ θα πρέπει να συνεχίσει να λειτουργεί αποτελεσματικά, θα χρειαστεί τα επόμενα χρόνια να στρέψει το βλέμμα της πέρα από τους παραδοσιακούς τομείς δράσης. Θα πρέπει να θετήσει μια, προοπτρο... μια προοπτική ε, επιτόπου σε συνεργασία και με τις εθνικές αρχές για να βρίσκεται όλο ένα και πιο κοντά στις ε, υγειονομικές ανάγκες των πολιτών και στα συστήματα περίθαλψης κοντά δηλαδή σε αυτούς τους θεσμούς, αυτούς τους φορείς που χειρίζονται την υγεία στην καθημερινή ζωή. Θα πρέπει να αναπτύξει μια ολιστική προσέγγιση για τη ρύθμιση των φαρμάκων και των φαρμακευτικών προϊόντων για να ε, συμπεριλάβει καλύτερα αυτό που μας δίνει η επιστήμη στις ε, ρυθμιστικές πρακτικές. Θα πρέπει να ενισχυθεί επίσης η συνεργασία στο εσωτερικό της, να ε, συνδυάσει, να συντονίσει καλύτερα τις δραστηριότητές τους αλλά και σε εξωτερικό επίπεδο γιατί ε, λόγω και έλλειψης πόρων ε, δεν θα μπορέσει ε, να προσφέρει την επαρκή προστασία στους ανθρώπους και στα ζώα. Βάσει της περασμένης, της παρελθούσας εμπειρίες μου και λόγω των διάφορων ευκαιριών που είχα ως επιστήμονας κινητρός και ως μάνατζερ, ως διευθυντής, νομίζω ότι μπορώ να συνεισφέρω στο EMA για να γίνει μια ενεργή δύναμη, η οποία θα παρέχει μια υγειονομική αρρωγή, οικονομικά προσβάσιμη και που θα βασίζεται στη διαφάνεια και στην ανεξαρτησία και την αμεροληψία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, για την ευκαιρία που μου δώσατε να παρευρεθώ εδώ και φυσικά Είμαι έτοιμος να απαντήσω στις ερωτήσεις σα και ελπίζω να σας απαντήσω και ικανοποιητικά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ράζη. Σας ευχαριστούμε για αυτό το όραμα περί της πολιτικής των φαρμάκων, ε, τι πολιτική πρέπει να ακολουθήσει ο οργανισμός τα επόμενα έτη. Σας ευχαριστώ ε, που σεβαστήκατε το χρόνο ομιλία σας και μάλιστα τα πήγατε και καλύτερα από αυτό που προτείνουμε εμείς. Έτσι λοιπόν, ε, θα πρότεινα για τον πρώτο γύρο να ξεκινήσουμε με την κυρία Γκροστέτη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Δευθυντά. υποψήφια Δευθυντά. Θα μιλήσω για μια υπόθεση που έχει ακουστεί πολύ στη Γαλλία. Πρόκειται για το σκάνδαλο των μεσολαβητών και ο Πίτροπος Δέλη ξεκίνησε, έθεσε εφαρμογή στρε τεστ για να δει αν τα νέα μέτρα φαρμακογρύπνησης που ψηφίσαμε πρόσφατα θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν και να εμποδίσουν ένα τέτοιο σκάνδαλο. Είδαμε ότι υπάρχουν ε, κάποια εύθραστα σημεία στην ομοθεσία μας για τη φαρμακογρύπνηση. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε τι προτίθεστε εσείς να κάνετε για να βελτιώσετε την κατάσταση και να λάβετε κάποιες ε, αποτελεσματικές αποφάσεις κατόπιν των αποτελεσμάτων των stress test. Και θέλω να σας πω τι σκοπεύετε να κάνετε για να λάβετε υπόψη τους κινδύνους που σχετίζονται ε, με τη χρήση ε, φαρμάκων για τους ασθενείς που είναι εκτός ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκου. Μάλιστα. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Τώρα δεν υπάρχει τεχνική λύση. Δεν έχω απάντηση. Παρακαλώ, αν θέλετε να απαντήσετε, έχετε το λόγο για δύο λεπτά, λεπτά κύριε Ράζη. Ναι, το πρόβλημα του μεσολαβητή είναι ένα θέμα που έχει συζητηθεί πάρα πολύ σε όλους τους οργανισμούς. Εγώ μπορώ να σας πω από τη σκοπιά της, ε, του Ιταλικού Οργανισμού προσπάθησα να παρακολουθήσω όλη αυτή την ιστορία του Μεσολαβητή, κατάλαβα ότι μία από τις μεγάλες αδυναμίες που υπήρχαν ε, στον, προηγούμενο νόμο της φαρμακοεπαγρύπνησης έχουν αντιμετωπιστεί, παραμένει να, μείνουν, να γίνουν με συγχωρείτε τα stress test και πρέπει να καλυφθούν κάποια κενά. Εγώ πιστεύω ότι Ευρωπαϊκό Οργανισμός Φαρμάκων καταρχήν θα πρέπει να εφαρμόσει τον νόμο και να συνδέσει τα εθνικά δίκτυα φαρμακοεπαγρύπνησης με το ενιαίο δίκτυο φαρμακοεπαγρύπνησης. Φυσικά η φαρμακοπαραγρύπνηση έχει και ένα άλλο κριτικό σημείο, τα σήματα, ε, τα μηνύματα της φαρμακοπαραγρύπνησης ε, πρέπει να είναι επαγγελματικά και εντελώ ε, σαφή. Η γλώσσα αυτής της φαρμακοπαγρύπνησης είναι επαγγελματικού χαρακτήρα. Η νέα νομοθεσία προβλέπει να υπάρχει και άμεση ε, πρόσβαση από τους ασθενείς και καταρχήν θα γίνουν κάποιες προσωμιώσεις για να δούμε ε, πόσο καθαρά είναι τα σήματα αυτά. Δεύτερο, να προσπαθήσουμε να εξορθολογήσουμε ε, τους πόρους όσο το δυνατόν περισσότερο γιατί θα μπορούσε να δημιουργηθεί κάποια σύγχυση βάσει αυτών των σημάτων. Ε, βάσει αυτών των καταγγελιών. Εγώ νομίζω ότι κατά τα λοιπά είναι εύρωστο το σύστημα και θα μπορέσει να καλύψει και κενά. Κύριε Γκροστέτ, ε, μιλήσατε για τον παιδιατρικό κανονισμό. Καλό είναι το ότι υπάρχει αυτός ο κανονισμός, όμως οι ερευνητές, ε, οι παιδίατροι λένε ότι δυσκολεύονται να εφαρμόσουν αυτόν τον κανονισμό ε, λόγω της διαχείρισης των κλινικών δοκιμών. Θα ήθελαν να έχουν λίγο μεγαλύτερη αυτονομία για το θέμα αυτό. Εσείς τι πιστεύετε. Παρακαλώ, κύριε Ράζη. Εγώ προφανώς ε, δεν θεωρώ ότι κατέχω τη λύση. Εγώ θέθετα την ερώτηση που μου κάνατε κι εσείς, δηλαδή με άλλα λόγια, είναι αλήθεια ε, να έχουμε ένα πείραμα, να γίνονται πειράματα για τα παιδιά, ε, πάνω στα παιδιά, κοιτάξτε, θέτει πραγματικά ηθικά προβλήματα, αλλά να μην το κάνουμε, παρουσιάζει και αυτό προβλήματα για την υγεία, για ορισμένα μελλοντικά ε, φάρμακα. Η επιστήμη πρέπει να μας δώσει νέους βιοδείκτες ε, και νέες ε, απαντήσεις σε κλινικό επίπεδο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποφύγουμε ένα μέρος του κινδύνου θα πρέπει φυσικά να αφήσουμε την τελευταία λέξη στους επιστήμονες, οι οποίοι αναπερίπτωση καθορίζουν τον αποδεκτό κίνδυνο για τα πειράματα, για ένα πείραμα. Δεν υπάρχει μία ενιαία λύση, θα πρέπει να τη βρίσκουμε ανάλογα με το φάρμακο και ανάλογα με την όσο που μελετάμε. Σας ευχαριστώ κύριε υποψήφια διευθυντά. Έχουμε και τον ε, ε, βουλευτή, ε, την κυρία που είναι σε επαφή με την EMA. Παρακαλώ. Ήθελα να ρωτήσω τον δόκτωρα Ράζη για μια πρωτοβουλία με την οποία ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα. Υπάρχει πάντοτε ο κίνδυνος να επισκιάσει η EMA, η EMA, τα, ε, το θέμα των ομοιοπαθητικών, α, των ε, φαρμάκων που προέρχονται από, φα, από φυτά, φυτικής προέλευσης. Είχα, έχω και περισσότερο καιρό γιατί ήμουν πολύ γρήγορη. Ήθελα να ρωτήσω λοιπόν τον δόκτωρ τον Ράζη ε, τι πιστεύει ότι μπορεί να κάνει για την πρόθεση των φαρμάκων με φυτική προέλευση. Και μια που έχω καιρό, να προσθέσω, να μου απαντήσετε στο πρώτο γύρο, αλλά μπορεί να με επικαλύψουν και άλλοι συνάδελφοι. Εάν έχετε κάτι να μας πείτε για τη σύγκρουση συμφερόντων με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Αξιολόγησης, τον Ευρωπαϊκό Φορέα Αξιολόγησης. Παρακαλώ, έχετε δύο λεπτά κύριε Ράζη. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα φάρμακα φοιτικής προέλευσης, εγώ νομίζω ότι η σημερινή νομοθεσία μας επιτρέπει να τα χειριστούμε με κατάλληλο τρόπο. Το κύριο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την, τον οργανισμό είναι ε, ότι έχουμε ένα επαρκή αριθμό μονογραφιών και παραμένουμε στην ίδια κατάσταση, έχουμε δηλαδή το ίδιο δυναμικό χωρίς να αυξάνεται η πόρη, ούτε η οικονομική πόρη, ούτε η ανθρώπινη πόρη, καθώς πρόκειται για διαδικασίες που δεν πληρώνονται Γι' αυτό το λόγο πολλά έθνη είναι κάπως διστακτικά να τα αναλάβουν. Θα μπορούσαμε λοιπόν να θέσουμε ότι κάθε δύο πληρωμένες διαδικασίες είναι υποχρεωτικό να έχουμε μία μη ε, πληρωμένη διαδικασία. Μία διαδικασία που δεν πληρώνεται. Δεν ξέρω πόσο θα είναι ικανοποιημένα τα κράτη-μέλη, όμως θα ήταν ε, μία αποδεκτή λύση. Κάθε δύο, κάθε τρει, τέλο πάντων θα το δούμε. Αυτό είναι ένα θέμα ισορροπία. Τώρα, αν κατάλαβα, με ρωτήσετε για κάτι για τη σύγκρουση συμφερόντων. Για το θέμα αυτό, Πιστεύω ότι το πρόβλημα έχει να κάνει με την διαχείριση. Δεν δηλαδή δεν αρκεί να κατεθέτει κανεί μια σελίδα με τι δηλώσει. Θα πρέπει συνεχίσει να γίνεται μια αξιολόγηση και να υπάρχει και διασταυρούμενος έλεγχος ε, με φαρμακολογικές περιπτώσεις. Ε, τουλάχιστον εγώ στο δικό μου οργανισμό φαρμάκων έκανα ένα τεστ και είδαμε ότι μπορούμε να αξιολογήσουμε τους εμπειρογνώμονες πρόκειται για μια δουλειά συνεχούς ε, αξιολόγησης. Ο οργανισμός ε, φυσικά δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά και μόνο, αλλά ένα έργο πιο προσεκτικό για την αναθεώρηση ε, μπορεί να γίνει διαφορετικά αν έχουμε ένα αποθετήριο που απλώς θα αποθέτουμε τις, ε, ε, τις αξιολογήσεις αυτές δεν φτάνει. Θέλω να επανέλθω στα φάρμακα φυτικής προέλευσης. Συμφωνείτε ότι χρειαζόμαστε περισσότερες μονογραφίες, χρειάζεστε ότι χρειαζόμαστε επίσης ε, και απλήρωτες αξιολογήσεις και πιστεύετε ότι όλο το σύστημα της έκδοσης και παρουσίασης μονογραφιών δεν λειτουργεί ε, ε, ικανοποιητικά και ότι χρειάζεται περαιτέρω εκπαίδευση στα κράτη-μέλη. Ο, ο κύριος και εκτελεστικό διευθυντή έχει το λόγο, υποψήφιο. Βεβαίως ε, μπορούμε να αυξήσουμε τη δέσμευση τη, EMA ε στο να ευνοεί αυτή τη συμμετοχή. Φυσικά υπάρχει μεγάλη ανεομοιογένεια στην επικράτεια της Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές αντιλήψεις. Δηλαδή η παραδοσιακή ιατρική είναι κάτι διαφορετικό, είναι το ένα, έχει ορισμένα συγκεκριμένα όρια. Ε, ε, όταν έχουμε μια ιατρική που προέρχεται από όλες υπήρους μπορεί να θέσει πρόβλημα. Εγώ πιστεύω ότι συμφωνούμε όλοι στο εξή, ότι πρέπει να έχουμε περισσότερη ασφάλεια σε σχέση με το τι διατίθεται στους ασθενείς κατά τα υπόλοιπα. Ε, ε, η νομοθεσία, αν εφαρμοστεί, ε, αρκεί. Όμως νομίζω ότι χρειάζεται μια προσπάθεια για την εφαρμογή της νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Μικρόφωνο για την Πρόεδρο. Λοιπόν, εγώ θα πάρω το λόγο εξ ονόματος της ομάδας μου. Λοιπόν, κύριε Υποψηφία, κλειστήκατε σε ένα άλλο ψήφισμα το 2011 θα επανέλθω στην ερώτηση του Ντάκμαρ ε, για τον προπολογισμό για το οικονομικό έτος ε, του 2009. Εμείς ε, είχαμε μία καταγγελία για τον προηγούμενο άτομο που εκτελούσε τα καθήκοντά σας. Είδαμε ότι είχε παραβιαστεί το άρθρο 6 του καταστατικού των υπαλλήλων. Χρειάστηκε να ασχοληθούν κάποιες μη κυβερνητικέ οργανώσει και κάποιες συναδελφοί μα, έτσι ώστε ε, τελικά ο ε, διευθυντής... Ε, να παρατηθεί και στο ίδιο ψήφισμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε στον εκτελεστικό διευθυντή του οργανισμού σε συνεργασία με τις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου να κάνει μια επαλήθευση βάθο για την ε, υφιστάμενη διαδικασία ταυτοποίηση και διαχείριση των ε, για τη σύγκρουση συμφερόντων. Τίποτα δεν γράψετε όμω εσεί στην επιστολή σα για το θέμα αυτό. Τι θα θέσετε σε εφαρμογή και ποιε πολιτικέ θα ακολουθήσετε σε σχέση με ε, την πρόσληψη των ατόμων αυτών αφού ε, θα έχουν περάσει από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Ma, devo dire che... Εντάξει, θα πρέπει να πω ότι στον προηγούμενο ρόλο μου ως ε, μέλος του Management Board ε, της ε, EMA και εμένα με προβλημάτισε εμείς στο Δικαιωτικό Συμβούλιο μάθαμε για την διαδικασία αυτή από τις εφημερίδες. Έτσι λοιπόν το Δικαιωτικό Συμβούλιο δεν ενημερώθηκε για το τι συνέβαινε. Και και νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα από τα πρώτα που θα κάνω, δηλαδή το Διοικητικό Συμβούλιο, θα φροντίσω το Διοικητικό Συμβούλιο να γνωρίζει όλα όσα συμβαίνουν στον οργανισμό και η σύγκρουση συμφερόντων είναι ένα από τα πλέον σημαντικά θέματα. Τώρα, εγώ δεν είμαι νομικός, έτσι λοιπόν δεν γνωρίζω ποιες είναι οι αρμοδιότητες του οργανισμού στο επόμενο στάδιο, όταν τελειώνει δηλαδή η θητεία ενός διευθυντή άλλων ε, ε, υπαλλήλων του οργανισμού. Βεβαίως και θεωρώ ότι το πρόβλημα αυτό είναι πολύ σοβαρό και θεωρώ ότι όσα γνωρίζει ένας υπάλληλος της CMA ε, μπορεί να είναι πληροφορία που θα τεθεί σε εμπορία εκτός και αυτό είναι ένα θέμα που μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Βέβαια ε, υπάρχει σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν πάλι που απλώς ε, ε, έχουν κάποιες γνώσεις και δεν ενδιαφέρουν οι γνώσεις αυτές τις εξωτερικές εταιρείες δεν ενδιαφέρονται δηλαδή να προσλάβουν το άτομο αυτό οι εξωτερικές εταιρείε. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να επαληθεύσουμε ποια είναι πραγματική νομική αρμοδιότητα ε, του οργανισμού και πιστεύω ότι το σωστό θα είναι όποιο αναλαμβάνει αυτά τα καθήκοντα να είναι πάρα πολύ προσεκτικός όταν ε, δέχεται στη συνέχεια ε, άλλα καθήκοντα, να λαμβάνει νέα καθήκοντα. Μάλιστα, πολύ σύντομα. Θα είμαι πιο σύντομη στην ε, επανάληψη ερώτησή μου. Λοιπόν, ε, καταρχήν ε, ε, στις συμβάσεις θα βάλετε συγκεκριμένους όρους για το όταν κάποιος αφήνει την εργασία του, αποχωρεί από την εργασία του. Και δεύτερον, θα αποκτήσετε κάποια μέσα ελέγχου των ενδείξεων που σας δίνονται. Δηλαδή, μιλάμε για κάτι πολύ συγκεκριμένο εδώ. Κοιτάξτε, το πρόβλημα των συμβατικών ρητρών. Ε, ναι, βέβαια, αν ε, υπάρχει δυνατότητα να το προβλέπουν οι κανονισμοί, ε, κοιτάξτε, αυτό το δέχομαι σαν ιδέα που μου λέτε εδώ, αλλά συμφωνώ. Θα μπορούσε να βρεθεί μια τέτοια λύση. Αυτό που επαναλαμβάνω ότι δεν ε, πρέπει να γίνει είναι να μετατραπούμε σε αστυνομικού. Σε αστυνομική δηλαδή πρέπει να υπάρχει έλεγχο, συνεχώ αλλά όχι να γίνει μια αστυνομική υπηρεσία. Και μία δήλωση σαφής ε, για το ποιος θα είναι ο ρόλος του ατόμου αυτού στα επόμενα καθήκοντα που θα αναλάβει είναι κάτι σημαντικό. Θα πρέπει να το δούμε βέβαια και σε συνδυασμό με το ότι χρειάζεται και κάποια προστασία. Ε, γιατί το άτομο αυτό, όπω και να έχει όταν θα αποχωρήσει από τον οργανισμό, θα πρέπει να βρει και μια άλλη δουλειά. Μάλιστα, ευχαριστώ κυρία Ριβάζη. Ευχαριστώ. Σε σχέση με την απάντησή σας, είμαι αρκετά ικανοποιημένη, γιατί όταν λέτε ότι το μάθατε από τον τύπο. Εγώ έχω εδώ την επίσημη απάντηση τη που λέει ότι ε, είχε εφαρμόσει αυστηρό του κανόνες. Έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά δηλαδή, αλλά θέλω να σας ε, κάνω μια ερώτηση για τα έγγραφα. Σύμφωνα με τη σημερινή πολιτική της ο έλεγχο ε, Επιτροπή τη της Φαρμακοκραγνύπνησης, οι ε, διαδικασίες αυτές δεν δημοσιεύονται όταν ολοκληρώνει τη διαδικασία. Το δικαστήριο έκρινε σε πολλέ περιπτώσει ότι αποτελεσματικότητα τη διαδικασία λήψη αποφάσεων για τα εσωτερικά έγγραφα δεν μπορεί να επικαλείται παρά περίπτωση και όταν η δημοσίευση των εσωτερικών εγγράφων συγκεκριμένα θέτει σε κίνδυνο τη διαδικασία λήψη αποφάσεων. Έτσι λοιπόν η EMA έκανε εξαίρεση για τον κανόνα. Θα ήθελα λοιπόν εγώ να μου πείτε, είστε έτοιμος να αλλάξετε αυτή την πολιτική του ΕΟΦ για να διασφαλίσετε ότι όλα τα πρακτικά θα γίνονται αυταπάγγελτα, θα δημοσιεύονται, δηλαδή να έχουμε πρόσβαση σε όλα τα πρακτικά που ε, αφορούν την συνεδρίαση της Επιτροπής Φαρμακοπαγρύπνησης και για τις κλινικές δοκιμές, για τα φάρμακα που θα τεθούν στην αγορά. Δηλαδή πρέπει να έχουμε διαφάνεια και διαφάνεια διαφάνεια περνά μέσα από τη δημοσίευση των πρακτικών των συνεδριάσεων και όλων των ε, κλινικών μελετών. Παρακαλώ. Κύριε Ναι, ευχαριστώ. Αλλά θα ξεκινήσω από το τελευταίο στο οποίο αναφερθήκατε, είναι το πιο εύκολο γιατί εκεί είμαι και σίγουρος για το τι σκεφτόμαι και για το τι είναι σωστό. Τα κλινικά δεδομένα, τα κλινικά στοιχεία πρέπει να δημοσιεύονται. Ήδη το κάνει η FDA και η EMA βέβαια στο θέμα αυτό έχει καθυστερήσει. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ε, για μη δημοσίευση μπορούμε να δούμε ποια είναι η στιγμή δημοσίευσης ορισμένων πραγμάτων αν αυτή η ενημέρωση μπορεί να ωφελήσει τη βιομηχανία, τον κλάδο, για να προσπαθήσει να επηρεάσει μια απόφαση που είναι ε, σε διαδικασία λήψης. Έτσι λοιπόν μπορούμε να αποφασίσουμε για τη στιγμή της δημοσίευσης. Όμως το ότι πρέπει όλα να δημοσιεύονται δεν έχω καμία αμφιβολία. Πρέπει να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να ξέρουν πώς ελήφθησαν οι αποφάσεις. Τώρα για το Διοικητικό Συμβούλιο, ας δούμε τις ημερομηνίε. Ευτυχώ έχω δύο λεπτά στη διάθεσή μου, λέει Λοιπόν, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημερώθηκε για τη διαδικασία αυτή αφού ε, είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία. Εμείς ε, δεν συμμετείχαμε στη συζήτηση πριν ε, να ληφθεί η απόφαση αυτή για τον πρώην εκτελεστικό διευθυντή. Εγώ προσωπικά στη συνέχεια δεν συμμετείχα στη συζήτηση που ακολούθησε γιατί ήδη ήμουν υποψήφιος για τη θέση του εκτελεστικού διευθυντή και θεωρούσα και αφού μας συμβούλευσε η Κοινωνική Υπηρεσία της CMA να μην κάνω δηλώσει γιατί θα μπορούσαν να ερμηνευτούν υπέρ ο κατά εμού δυνάμει και τη ε, υποψηφιότητάς μου. Μάλιστα, ευχαριστώ κυρία Ριβάζη για 30 δευτερόλεπτα. Ναι. Κοιτάξτε, δεν μου απαντήσατε για τα πρακτικά των συνεδριάσεων τη Επιτροπή Φαρμακοπραγνύπνηση. Και τελευταία ερώτηση για τι ανεξάρτητε και διαφανεί κλινικέ έρευνε. Σύμφωνα με πληροφορίε που είχα ω ε, ε, Γενικό Διευθυντή ε, του Ιταλικού Οργανισμού Φαρμάκων, δεσμευτήκατε κατά τη ανεξάρτητη κλινική έρευνα στην Ιταλία. Έτσι λοιπόν, ποια είναι η θέση σα για την ανεξάρτητη κλινική έρευνα μπορείτε να δεσμευτείτε ότι θα δημοσιεύει όλα τα στοιχεία ε, για την ιδιωτική αλλά και τη δημόσια κλινική έρευνα. Παρακαλώ κύριε Διευθυντά, κύριε υποψήφιε Διευθυντά. Κοιτάξτε, σε ό,τι αφορά τη συνεδρία τη Επιτροπή Φάρμακο Επεραγρύπνηση, ε, εγώ σκοπεύω να καταστήσω δημόσια όλη τη διαδικασία, φυσικά και τη συνεδρία της SMP ε, από τη στιγμή που δεν επηρεάζεται ε, το αποτέλεσμα. Τώρα, για την κλινική ερευνά, εγώ το πρόθεσα στην Ιταλία, έχουμε 180 μελέτες που ε, χρηματοδοτούνται η βάση επενδύσεων που έγιναν το 2004 στο 2010 δεν είχαμε ακόμη κανένα αποτέλεσμα και πήραμε τους πόρους και τους επενδύσαμε σε νέες κλινικές μελέτες. Τώρα 56 abstract είναι υποδημοσίευση με, με ε, περίπου 50 ε, σημεία για παράγοντες αντικτύπου. Σας ευχαριστώ. για την κουέ, Δεν υπάρχει κανείς, μάλιστα. Να δώσω το λόγο στον κύριο Πίτερ Λίζε για το δεύτερο γύρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε υποψήφιε, εκτελεστικέ διευθυντά. Έχω ένα θέμα για την νομοθεσία για τις ε, προηγμένες θεραπείες, ε, advanced therapies μετά από μακροχρόνιες ε, διαβουλεύσεις ε, πέντε ετών ε, φτάσαμε στο, από το 2007 είμαστε τώρα στο 2011 και σε αυτό το διάστημα μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας ένα προϊόν όμως έχει μόνο έχει αδειοδοτηθεί Ρωτώ λοιπόν αν αυτό είναι πρόβλημα της νομοθεσίας. Έχω ακούσει και από εταιρείε οι οποίες έχουν υποβαθμίσει ε, διάφορες ε, θεραπείες. Άρα λοιπόν η διαδικασία είναι πάρα πολύ γραφειοκρατική. Μήπως ξέρετε πώς μπορούμε αυτές τις προηγμένες θεραπείες να τις ε, υποστηρίξουμε έτσι ώστε να εφαρμόζεται σωστά η νομοθεσία. Κύριε Διευθυντή, υποψήφιε Διευθυντά, έχετε το λόγο. Κοιτάξτε, είναι πρόβλημα νομοθεσία. Ναι, κοιτάξτε, η ΕΜΕ έχει μια μεγαλύτερη επιρροή για την ενημέρωση. Εγώ πιστεύω ότι είναι πρόβλημα νομοθεσία, όπω ε, είπατε. Ε, κάθε πέντε χρόνια δίνεται άδεια σε ένα φάρμακο. Και τι γίνεται ε, κάποιες εταιρείε προσπαθούν ε, να περάσουν αυτές τις προηγμένες ε, θεραπείες της advanced therapies ως θεραπείες στο νοσοκομείο, σε τοπικό επίπεδο ή με κάτι που να μοιάζει με τα device, με τις συσκευές. Δηλαδή προσπαθούν να ακολουθήσουν μια πιο απλή νομοθεσία. Αυτό δεν είναι καλό ούτε για τις επενδύσεις, ούτε για τους ασθενείς, ούτε για την ανάπτυξη φαρμάκων που μπορεί να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και αποτελεσματικά θα πρέπει εδώ να δεχτούμε ότι αυτή η νομοθεσία τελικά δεν πληρεί τους σκοπούς της. Έχουμε ένα μεγάλο μηχανισμό ετών και προσπαθειών ε, που τελικά κατέληξαν σε αυτό που είπατε εσείς. Είναι προφανές. Δεν το αμφισβητούμε. Κοιτάξτε, προσωπικά εμένα με ενδιαφέρει πολύ αυτό το θέμα, γιατί στην προηγούμενη ζωή μου, όταν ήμουν επιστήμονας, ασχολούμουν ε, ακριβώ με αυτές τις θεραπείες. Έτσι λοιπόν με ενδιαφέρει πάρα πολύ να αναπτυχθεί κάτι τέτοιο, γιατί η δυναμική θεραπεία που έχουν αυτές οι τεχνολογίες είναι τεράστια. Σίγουρα πρέπει να ξαναδούμε και το θέμα της γραφειοκρατίας. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και νομίζω ότι αυτή είναι η έδρα όπου πρέπει να θέτουμε τα προβλήματα και θα πρέπει να δούμε πώς θα προκύψουν και οι λύσεις να σας ρωτήσω εκ μέρους ε, των διερμηνών που με λίγο από το μικρόφωνο, λέει η Πρόεδρος. Μάλιστα, δικαίωμα απάντηση σε ένα λεπτό. Έχετε. Ναι, μια συμπληρωματική ερώτηση. Πρέπει να συνεργαστούμε να δούμε τι μπορεί να γίνει χωρίς αλλαγή της νομοθεσίας, τι μπορεί να βελτιωθεί σε επίπεδο ΕΟΦ. Το Κοινοβούλιο έχει προτείνει να γίνει εκ νέου επεξεργασία της νομοθεσίας. 2009 αρχίζει η σύμβαση διανομής όπου γίνεται υποχρεωτική η μη εμπορευματοποίηση του ανθρώπινου σώματος ή μερών του ανθρωπίνου σώματος. Φαντάζομαι ότι αυτό πρέπει να ισχύσει και για ιστούς και για κύτταρα. Και αν χρειάζεται η προσαρμογή της νομοθεσίας πρέπει να γίνει και σε αυτό, δεδομένου ότι ισχύει πλέον αυτή η σύμβαση. Κύριε Δευθυντά, υποψήφι. Προσωπικά Πιστεύω ότι η δεν είναι, θέση σε εμπορία δεν είναι κάτι κατάλληλο. Μπορούμε να έχουμε παράβλεπες δαπάνες, αλλά δεν νομίζω ότι ο ίδιος ο ανθρώπινος ιστός θα πρέπει να είναι αντικείμενο εμπορίως. Στη νομοθεσία, στη χω... βάση της νομοθεσίας της χώρας μου μπορεί να δώσει κάποιο αίμα μόνο εθελοντικά και νομίζω ότι είναι καλή η προσέγγιση αυτή. Μικρόφωνο παρακαλώ για την Πρόεδρο. Ευχαριστώ. Να δώσω τώρα το λόγο. Συνάδελφο Λίντα Μακαβάν δεν είναι εδώ. Όχι εδώ είναι. Μάλιστα. Λίντα Μακαβάν. Άλλαξα. Άλλαξα γιατί δεν ακούω καλά από εκεί που καθόμουν. Λοιπόν, αναφέρεται ότι υπάρχουν πολλές νέες προκλήσεις σε αυτόν τον αιώνα και πολλά πράγματα θα αλλάξουν. Μπορείτε να μας πείτε τι εμπειρία έχετε από τη διαχείριση μεγάλων αλλαγών σε έναν οργανισμό. Παραδείγματος χάρη μπορείτε να μας δώσετε παραδείγματα μεγάλων αλλαγών τα οποία εφαρμόσατε ή διαχειριστήκατε σε οργανισμούς στους οποίους εργαστήκατε. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, φέρνει σε δύσκολη θέση αυτή η ερώτηση γιατί ειναι μιλάει κάποιο για κάτι που θεωρείται είναι επιτυχία, μπορεί οι άλλοι να μην συμφωνούν. Ε, εγώ έκανα δύο μεγάλες αλλαγές ε, στον οργανισμό. Άλλαξα το σύστημα διακυβέρνησης, ε, governance, το σύστημα διαχείρισης αυτή τη στιγμή όπου υπήρχε περιορισμός στις προσλήψεις προσωπικού. Από 250 όμως ε, φτάσαμε στα 500 άτομα. Στα πλαίσια του ίδιου προπολογισμού εξορθολόγησα λοιπόν ε, επαρκώς τις διαδικασίες και τις δραστηριότητες. Και ε, προώθησα την ανεξάρτητη έρευνα γιατί αυτό ήταν το background του μου, αλλά τη μετέτρεψα σε μία έρευνα που ουσιαστικά είχε να κάνει με αποφάσεις για το πώς διαχειριζόμαστε τα φάρμακα και ε, με το τι γίνεται με τη συνταγογράφηση των φαρμάκων. Ε, επίσης, μιλούσα τρεις σημαντικά ε, τρεις σημαντικές τράπεζες παιδιατρίας για τους ηλικιωμένους και για την παθολογία, για τη γενική ιατρική. Μια άλλη πτυχή ήταν ε, ότι προσπάθησα να ε, προσδώσω στον οργανισμό στην Ελλάδα μεγαλύτερη ανεξαρτησία απέναντι στη βιομηχανία κυρίω. Δημιουργήσαμε μια βάση δεδομένων εμπειρογνωμόνων και ζητήσαμε από τις εταιρείε να μας δώσουν τη δική τους, ε, τις δικές τους βάσεις δεδομένων και κάναμε διασταυρούμενο έλεγχο και είχαμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Βέβαια, εν μεταξύ, ε, πέρασε ο καιρός και έληξαν αυτά τα στοιχεία. Λοιπόν, αν θέλετε και λίγο περισσότερο χρόνο, νομίζω ότι δεν υπάρχει... Γιατί έληξε ο χρόνο, υπομιλητή και λέει ο πρόεδρο, «Ε, έχετε περισσότερο χρόνο αν θέλετε, δεν θα υπάρχει αντίρρηση. Παρακαλώ, Λίντα. Προτιμώ να τελειώσει αυτό το οποίο έλεγε ο κύριος εκτελεστικός διευθυντή, υποψήφιος. Γιατί βεβαίω το ένα είναι να διοικεί και το άλλο είναι να φροντίζει να συμβαίνουν πράγματα και να αλλάζει το σύστημα. Ξέρω πως η Κομισιόν ε, τυπικά είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της νομοθεσίας. Στην πραγματικότητα, εάν δεν προωθήσει την αλλαγή υπηρεσία, δεν θα γίνει αυτό. Γι' αυτό θέλω ε, και έκανα αυτό το ερώτημα. Ε, ε αν ε, μιλάτε για την εμπειρία μου στον τελικό οργανισμό, οι διάφορες αποφάσεις ε, που ελήφθησαν, παραδείγματο χάρη το, για την νομοθεσία, για τη ρυθμίση των ορφανών φαρμάκων, για τους τρόπους πρόσβασης, Εμείς ε, κατορθώσαμε να αλλάξουμε τις ε, πρακτικές και μπορέσαμε τελικά να δημιουργήσουμε ένα οργανισμό που να σέβεται τα ευρωπαϊκά πρότυπα και επίσης ε, λάβαμε και την έγκριση της ΜΠΕΜΑ και πήγαν αρκετά καλά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, όπως βλέπετε, μετατράπηκαν όλα αυτά σε μια δράση και ε, οδηγήσαμε τον οργανισμό στο να έχει πάρα πολύ καλές επιδόσεις. Είναι δύσκολο να μιλήσουμε για τις επιτυχίες κάποιου. Ξέρετε τώρα, το, κάτι πολύ σημαντικό που άλλαξε την οτροπία του οργανισμού μου, που είναι το ότι ε, πέρασε ε, από την εξής νοοτροπία στο ότι παρέχει μία υπηρεσία, σε μια υπηρεσία που τη οποία κάθε δράση έχει άμεση επίπτωση στην υγεία των πολιτών. Γιατί δεν πρόκειται πλέον για καθήκον. Ευχαριστώ τον κύριο Ζήπερ τώρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε υποψήφιοι εκτελεστή και διευθυντή. Υπάρχουν τέσσερις διαδικασίες έγκρισης νέων φαρμάκων. Διαπιστώνουμε πως τα τελευταία χρόνια ακολουθούμε μια κεντρική διαδικασία πολύ περισσότερο. Αυτό σημαίνει βεβαίως πως και η δουλειά του ΕΟΦ γίνεται πολύ μεγαλύτερη. Όσον αφορά δε, και το προσωπικό σας, πώς κρίνετε ε, ότι θα μπορέσει να διατηρήσει την ποιότητα των γνωμοδοτήσεών του και ποια μέτρα θα θέλατε να λάβετε για την ανταγωνιστικότητα που αναφέρατε και εσείς της Ευρωπαϊκής Φαρμακοβιομηχανίας, γιατί είναι ένα βασικό θέμα του πώς ε, θα μπορέσει να προοδεύσει η Ευρωπαϊκή Κοινωνία. Ε, Ακούστε, Καταλαβαίνω τι γίνεται. Νομίζω ότι είναι η εξοδότηση για να κυκλοφορήσει το φάρμακο, γιατί στον όφο ακριβώ ε, αυτό κάνουμε. Δεν ξέρω μήπως εγώ δεν κατάλαβα σωστά. Η όλη διαδικασία για την χώριση άδεια θα μπορούσε να αλλάξει πραγματικά αυτό που συμφωνείται και η πρώτη προσέγγιση ώστε να αλλάξει ιδιαίτερα η όλη ταχύτητα απόφασης είναι η αποτελεσματικότητα του Scientific Advice να αλλάξει προς το καλύτερο. Όσο γίνεται νωρίτερα αυτό με το ίδρυμα που θέλει να αναπτύξει ένα φάρμακο τόσο όσο έχουμε καλύτερους κοινού δρόμους, τότε πιο πιο εύκολο θα είναι να προχωρήσει όπως είναι η πρόβλεψη για το φάρμακο. Βέβαια η βιομηχανία δεν μπορεί να αντέξει μια βεβαιότητα. Αυτό το αμερικανικό παράδειγμα θα μπορούσε σε μερικές περιπτώσεις να εφαρμοστεί και με μια άμεση επαφή πολύ πολύ γοργή προκαταρτικά με τη βιομηχανία και πολύ συχνά αυτό το trial, τα κλινικά, τις κλινικές δοκιμές ε, όπως έχουμε συμφωνήσει με τις ΗΠΑ και που γίνονται δεκτοί και από τον ευρωπαϊκό πληθυσμό. Εδώ στο ξεκίνημα μπορούν να παιχτεί όλο το παιχνίδι για την βελτίωση αποτελεσματικότητα του συστήματο. Και ακόμα ένα πρόβλημα σχετικά πάντα με το scientific advice. Ε, σημαντικό είναι κατά την απόψή μου να μπορέσουμε να συνδυάσουμε και το technology assessment, αυτή τη διαδικασία, για να αποφύγουμε ακριβώς, ε, για να δώσουμε μια άδεια ε, για ένα φάρμακο που κανείς δεν θέλει μετά να πληρώσει τη χορήγησή του. Αυτό, πάνω σε αυτό θα πρέπει να προχωρήσουμε πιο σύντομα, πιο γρήγορα και με καινοτόμε ε, λύσεις που θα συμμερίζονται όλοι. Κύριε Ζήμπερ. Τι μπορούμε να κάνουμε ε, για να γίνουν πραγματικά πιο φτηνά τα φάρμακα. Υπάρχουν πάρα πολλά ακριβά φάρμακα και αναφέρατε εσείς ακριβώς ότι πρέπει να έχουν προσιτές τιμές. Τι θα κάνει ο ΕΟΦ για αυτό το πράγμα. Eh, ο ΕΟΦ δεν συμμετέχει στη διαδικασία αυτού του ορισμού τιμής ε, του φαρμάκου. θα πρέπει οι διάφορες ρυθμίσεις σχετικά με την ε, άδεια κυκλοφορία θα πρέπει να λειτουργήσουν όπως πρέπει και να μειωθεί το κόστος στη βιομηχανία κλπ. και έτσι να μειωθεί γενικά και το τελικό κόστος του φαρμάκου. Το να γνωρίζει κανείς ε, το HTA τι θα γίνει εκεί. Και αυτό μπορεί να παίξει ρόλο στη μείωση του κόστους επένδυσης και τελικά θα πρέπει να είναι μια μείωση του κόστους και καλύτερη πρόσβαση. Θα πρέπει όλα αυτά να γίνονται βέβαια με ασφαλή τρόπο και η ευχή μου είναι να μας βοηθήσει και επιστήμη με νέα in-point κλινικά που να μην κοστίζουν. Α, λοιπόν, να επαναδιαγραφεί αυτό περί κλινικού πειραματισμού και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την διαδικασία στη συνέχεια. Σας ευχαριστώ. Ζηλ Παρνιό τώρα. Δύο λεπτά. Μάλλον ένα το. Ευχαριστούμε τον Διευθυντή. Θα ήθελα τώρα εδώ να έλθω στο θέμα των ε, συνταγών εκτός από του συστήματος αυτού όπως το είπε η κυρία Γκροστέτ πριν από λίγο. Η RMM είναι 15% με 20% των ε, συνταγών σε ηριατρία, καρκινολογία, παιδιατρία και το είδαμε τώρα τελευταία. Αυτό δημιουργεί και ένα κάποιο φόβο μπορούμε να πούμε από αρκετούς ε, συμπολίτες μας εργοστάσιο Pfizer για τον ερωτάν, για το φάρμακο που ήταν κατά της επιλεψίας και θα ήθελα να βοηθήσει διάφορες διπλής κατεύθυνσης εκδηλώσεις νευρολογικές και εδώ εσείς τι θέλετε να υιοθετήσετε για να πετύχετε μια καλύτερη διαφήνεια, φάνεια σχετικά με αυτή τη χρήση εκτός IMM και τι επιθυμείτε έτσι να λάβετε μέτρα για μια άμεση αποτελεσματική απάντηση και ανταπόκριση σχετικά με αυτούς τους φόβους και τις ανησυχίες που δημιουργούν οι χορηγείς φαρμάκου εκτός του συστήματος αυτού αρκε... υψηλού αριθμού φαρμάκων. Ναι. Ακούστε, το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό το φλεβελ το σύστημα περί φαρμάκων και στην παιδιατρική αποτελεί κανόνα μάλλον παραεξαίρεση ακριβώς ε, είπαμε για, τις κλινικ, τα κλινικά τεστ που δεν περιλαμβάνουν όμως παιδιά σας τη διαδικασία. Το Ίδρυμα τώρα κατά πόσο θα μπορούσε να περάσει την κατάσταση δεν γνωρίζω, δεν ξέρω. Αν υπάρχει ένα περιθώριο θα το κάνω χρήση του και το Ίδρυμα μήπως θα μπορούσε να το κάνει μαζί με την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο, στην συνεργασία μαζί τους. Αλλά ο ΕΟΦΕΞ ε, ξορισμού καθορίζει το on-level και αυτό που, για το οποίο δίνουμε άδεια εμείς είναι αντίθετο με αυτό που λέω και παρόμοιες δραστηριότητες ε, ελέγχου επαγρύπνησης ε, έχει να κάνει με χίλιες δυο φορείς ε, περιφερειακούς εθνικούς και έχει να κάνει και στο τέλος αλυσίδας με τον μεμονωμένο γιατρό. Ακριβώς αυτό για τις ε, συνταγές. Όλα αυτά δεν είναι μόνο από τη ρυθμιστικό ίδρυμα που καθορίζεται. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε εάν οτιδήποτε συντονισμένο θα μπορούσαμε να το αποδεχτούμε που θα γίνει προς την κατεύθυνση αυτή. Τώρα όσον αφορά τις προτάσεις, ε, εκείνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι από πολιτιστική σχεδόν πλευράς ε, κάτι το ιδιαίτερο, να προωθήσουμε κατευθυντήριες γραμμές και να έχουμε στη διάθεσή μας και τη νομική βάση, ώστε αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές να, είναι, ε, να μπορούν να λειτουργήσουν, να εφαρμοστούν και να υπάρχει μια κωδικοποίηση του φαρμάκου περισσότερη καλύτερη. Και κάθε νέα ένδειξη σε ένα φάρμακο βλέπουμε ότι από την χρήση του φλέμπελ έτσι ε, φαίνεται σε όλη του την έκταση. Και το συλφαμιδούργια για, τους διαβητικούς, τα συλφαμιδικά ακριβώς από που προήλθαν ε, χρησιμοποιώντας σουλφαμιδικό για μολύνσεις, έτσι, και ήταν ε, παρενέργεια. Και είναι, μπορούμε να πούμε, και πολιτιστικό, ας το αποκαλέσουμε έτσι θέμα και μάλιστα πολύ σημαντικό. Κύριε Παρνιό, δεύτερο ερώτημα ακριβώ. Ε, και μετά από την απάντησή σα και μετά από όσα είπε η κυρία συντονίστρια. Εσείς, ε, διευθυντή του ΕΟΦ, που να τα παροτρύνετε τα αριστερά φαρμακευτικά στη χρήση αυτή εκτός RMM να μπορέσουν να κάνουν και πάλι μια εκτίμηση των φαρμάκων ε, όπου δεν είχαμε διάφορες ιδιότητες, ε, κυρίως τις πληροφορίες που οι υπηρεσίες καταγραφής έχουν δει και ακριβώ τι μπορείτε να κάνετε. Ακούστε. Ο ΕΟΦ κατά την απόψή μου θα μπορούσε να επηρεάσει ιδιαίτερα έτσι, τις απόψεις, την φιλοσοφία και, την, και επιστημονικά επίσης. Όταν ε, φάρμακο χρησιμοποιείται κατά τον τρόπο αυτό, έχει αποδειχτεί ότι θα μπορούσε να βοηθήσει και ο ΕΟΦ ε, θα μπορούσε μια αγοργή ανείχνευση να οργανώσει και να μειώσει όσο γίνεται τις ε, επενδύσεις, αλλά βέβαια τις ελάχιστες τουλάχιστον για μια ασφάλεια για να δούμε νέες ενδείξεις που εμφανίζονται όμως σύμφωνα με τα όσα συνήθως ισχύουν για την άδεια κυκλοφορία χωρί κλπ. Λοιπόν, μια αγοργή ανείχνευση θα αποτελούσε μια καλή λύση, αλλά χρειάζεται να το δούμε αυτό, εάν πρόκειται ακριβώ για την προσέγγιση και μάλιστα τη σωστή. Σας ευχαριστούμε κύριε Διευθύντα. Το λόγο έχει ο Κιστανότ. Ε, σας παρακαλώ αφήστε να μιλήσει ο επόμενος ομιλητής από το ΕΛΚΟ, ο κ. Μπαρτολότσι νομίζω. Κύριε Διευθυντά, σας ευχαριστούμε. Κάτι να σας ρωτήσω. Το σύστημα φαρμακοεπαγρύψης, πώς να τον ισχύσετε για ένα έλεγχο των τοξικών ε, παρενεργειών μετά από την κυκλοφορία στην αγορά. Τι ακριβώς, ε, με ποιες πρωτοβουλίες θέλετε να ενισχύσετε εσείς ε, αυτή την αντιμετώπιση. Ε, εδώ λοιπόν. θα ήθελα Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Και επανερχόμαστε έτσι στην φαρμακοεπαγρύπνηση. Σας το είχα πει αρχικά πρόβλημα, θέμα πώς θα συνδυάσουμε τοπικές συνήθειες σε εθνικό επίπεδο και το entra vigilance όπως αποκαλείται εδώ αποτελεί ένα πρόβλημα και μάλιστα μεγάλο ποιοτική εμφάνιση ενδείξεων. Θα πρέπει αυτό το network που έχει ο ΕΦ και που το χρησιμοποιεί όλα και περισσότερο μάλιστα το ICM και για, τους, για τα στελέχη ακριβώς του Ιδρύματος για να δει πώς θα μπορούσαμε όσο γίνεται ταχύτερα να συνδυάσουμε τα τοπικά συστήματα φαρμακοκορύμψης με το κεντρικό σύστημα. Βέβαια και έχουμε παράπλευρες ενδείξεις ε, και με την οδηγία αυτή περί φαρμακοεπαγρύπνησης για την οποία αναφερθήκαμε με μια σειρά post-marketing ε, ε, ζωτική σημασία ενδείξει από τα διάφορα μητρώα στα ευρωπαϊκά κράτη και έτσι μάλιστα με επιλεκτικό τρόπο να δουν διάφορα στοιχεία για φάρμακα που με είναι ιδιαίτερα σοβαρά, ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και έτσι να δούμε αυτές τις ενδείξεις, να δούμε την επεξεργασία του, την αποκρυπτογράφησή του κατά κάποιο τρόπο και να μα δώσουν πληροφορίε και μάλιστα πολύ πιο γρήγορα πάνω σε τόσο σημαντικά γράμματα, ε, φάρμακα και έτσι να έχουμε μείωση του κόστους χωρίς ιδιαίτερες προσπάθειες, απλά και μόνο να δούμε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία ακριβώ που υπάρχουν ήδη. Ναι, ευχαριστούμε. Να πούμε, ο κ. Μπαρτολότσι για να πει ακόμα μερικά πραγματάκια, συμπληρώνοντας, ακούστε, τι θέλω να ρωτήσω. Σχετικά με αυτό που εσείς περιγράψατε και θέλετε να προωθήσετε η σημερινή νομοθεσία και η ευρωπαϊκή βέβαια και η μονομένα εθνική ε, σέβονται όλα αυτά σύμφωνα με την ε, επιδίωξη αποτελεσματικότητα των στόχων για την φαρμακοϊπαγνύπνηση την οποία αναφέρατε. Όπω έχουν τώρα οι νόμοι για τη φαρμακοεπαγρύπνηση, η ευρωπαϊκή σίγουρα είναι και περισσότερο προχωρημένη το stress test έδειξε και ορισμένες αδυναμίες που θα μπορούσαν ίσως να αποτελέσουν αντικείμενο μιας κάποιας τροποποίησης, αλλαγής και που έχει γίνει και σε τοπικό επίπεδο ο πλευρά ΕΟΦ. Τώρα το αδύναμο σημείο στην υπόθεση είναι ότι όταν αποσύρεται τις κυκλοφορίες από μια χώρα και μας για λόγους ασφάλειας το φαρμακό θα πρέπει οπωσδήποτε να ενημερωθούν και οι υπόλοιποι και να αποσυρθεί και σε όλα τα κράτη έτσι να μπορούν να αντιδράσουν ανάλογα είτε και να γίνει κάτι το υποχρεωτικής φύσης για τον ΕΟΦ και να υποδείξεις ε, όλων το, όλα τα κράτη την απόσυρση. Εκεί όμως είναι και το αδύναμο σημείο. Ευχαριστώ. Ο κ ήρθε εδώ και για ένα λεπτουδάκι να μας πει κάτι. Ευχαριστώ, εδώ ήμουνα, αλλά δεν περίμενα τόσο γρήγορα να μιλήσω. Μιλήσατε ήδη για το θέμα της διαθεσιμότητας των φαρμάκων και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ξέρετε πως έχουμε δύο διαδικασίες αδειοδότησης, μία κεντρική και μία εθνική και όταν ε, μιλάμε με τους ερευνητές ε, και τις φαρμακοβιομηχανίες παραπονιούνται συνέχεια για την πολυγραφειοκρατία, το κόστος ε, σε σχέση με αλλού. Και επειδή υπάρχει αυτό το κόστος δεν υιοθετούν την κεντρική διαδικασία και βεβαίως η άλλη διαδικασία οδηγεί στο ότι ζητάνε και άλλες διαδικασίες σε άλλες χώρες. Ο ΕΟΦ λοιπόν θα μπορούσε να έχει μια τυποποιημένη διαδικασία που θα ισχύει πανευρωπαϊκά και για εθνική αδειοδότηση και έτσι να μειωθεί το κόστος και η γραφειοκρατία. Και νομίζω θα βελτιωθεί και η κατάσταση όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των φαρμάκων. Το ερώτημά μου είναι λοιπόν εάν συμφωνείτε με μια τέτοια ερμηνεία ή εάν λέτε πως δεν μπορεί να εφαρμοστεί κάτι τέτοιο. Το δεύτερο ερώτημα αφορά την ε, αντοχή, την αντοχή στα αντιβιωτικά. Είναι πολύ σημαντικό θέμα τελευταία. Έχουν τεθεί πολλά ερωτήματα και η Επιτροπή Γεωργίας του Κοινοβουλίου ενέκρινε ένα ψήφισμα που αναφέρει πάρα πολλά θέματα και υποβάλλει πολλές προτάσεις ε, που πρέπει και να εφαρμοστούν. Όσον αφορά λοιπόν την αδειοδότηση των αντιβιωτικών, θα μπορούσατε να έχετε μια άλλη διαδικασία που θα αφορά ειδικά το θέμα της αντίστασης στα αντιβιωτικά για να υπάρξει και καλύτερη ε, εφαρμογή ως προς αυτό όσον αφορά την ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά. Ε, ναι, για την, την ιατρική νομοθεσία Σίγουρα υπάρχει ένα πρόβλημα και μάλιστα σημαντικό γραφειοκρατίας. Η πρότασή σας, ε, την πρότασή σα μπορούμε να τη συμμεριστούμε για να θέσουμε σε κεντρικό επίπεδο και να είμαστε όσο γίνεται περισσότερο υπέρ μια εναρμόνιση στα ευρωπαϊκά κράτη. Τώρα για τα κτηνιατρικά ξέρουμε τη δυσκολία πρόσβασης και μελέτης και για μικρότερα είδη που εκπροσωπούνται ελάχιστα. Κατά την άποψή μου το πρόβλημα αυτό σε κεντρικό επίπεδο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από τον ΕΟΦ και συμφωνώ από αυτού. Για την αντίσταση στα αντιβιωτικά, δύσκολο είναι να ξέρουμε η σωστή παρέμβαση ποια θα είναι, ποια είναι και να δούμε τη μηχανία που κάνει επενδύσεις πάνω σε αυτό. Δεν έχουμε πια καινούρια μόρια, καινούριε ουσίε και υπάρχουν 4-5 ουσίες μόνο, φόρμουλες που θα μπορούσαν να υποσχεθούν επιτυχία για το μέλλον. Να σα πω τίμια τίμια ότι η σωστή νομοθετική απόφαση ποια θα ήταν δεν θα ξέρα. Σίγουρα χρειάζεται να δούμε αυτή τη νομοθετική ε, διαδικασία, κάτι που ενθαρρύνει τη βιομηχανία στον τομέα αυτό να επενδύσει, αλλά ταυτόχρονα να περιορίσει την χρήση των αντιβιωτικών. Και επαναρχόμαστε έτσι στο προηγούμενο, στο φλέμπελ, στη χρήση αυτή, όπως είχε ζητήσει η συνάδελφος. Θα πρέπει ίσως να δούμε και κατευθυντές γραμμές, έστω και ένα δικό μας χρέος να λέμε στο γιατρό τι πρέπει να κάνει. Αλλά αυτές οι κατευθυντές γραμμές μερικές φορές να αποτελούν κάτι το υποχρεωτικό δεσμευτικό και αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει και στην ξέρεση πάνω στην οποία μπορούν να γίνουν τα πράγματα. Σας ευχαριστώ. Τώρα ναι. Δεύτερο ερώτημα το υποβάλλατε. Ναι. Ο Βιτόριο Πρόεδρε έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο καθηγητή, τον ευχαριστώ που είναι εδώ ανάμεσά μας. Θα ήθελα να αναφέρω μερικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη βακτηριοαντίσταση των, στα αντιβιωτικά. Και μετά από μια συζήτηση πριν από κάνα δύο εβδομάδες στο Κοινοβούλιο με το Γενικό Διευθυντή από τα κύριε ε, σημαντικότερα εργαστήρια τα φαρμακευτικά στον κόσμο και έλεγε ότι δεν ασκείται πίεση πραγματική για τη μελέτη νέων φαρμάκων. Αυτά τα κέρδη που θα μπορούσε να πετύχει με τα αντιβιωτικά είναι ελάχιστα. Τι μου ανέφερε σαν παράδειγμα μια κάποια αλλαγή κατεύθυνσης ε, της έρευνας προς ε, σπάνιες ασθένειες ε, με ένα φάρμακο ας πούμε για τον καρκίνο του προστάτη που κοστίζει όμως πολλά χρήματα έστω και αν είναι μόνο προς όφελος ελαχίστων ασθενών αλλά κοστίζει δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε όλο τον κύκλο χορήγησης. Θα πρέπει να δούμε σφαιρικά το πρόβλημα κατά την απόψή μου. Να πετύχουμε δηλαδή μια νέα ισορροπία και να έχουμε έτσι την εγγύηση ότι σε κάθε πτυχή της έρευνας θα καλύπτεται από την φαρμακομηχανία και να ρίχνει και μια ματιά στο θέμα της βασικής έρευνας στην ανάπτυξη αυτών των φαρμάκων που διευκολύνουν κατά κάποιο τρόπο τις δραστηριότητες αυτές ε, της έρευνας. Και ε, έχετε το λόγο κύριε Διευθυντά, χωρίς μικρόφωνο. Λοιπόν, το πρόβλημα αυτό της ε, αντίστασης των βακτηριδίων στα αντιβιωτικά σίγουρα έχει να κάνει και με τα νέα φάρμακα αλλά και τη χρήση των σημερινών. Και το δεύτερο θέμα, τη χρησιμοποίηση των σημερινών φαρμάκων που είναι ακόμα δραστικά και τα έχουμε στη διαθέσή μας πάντα, θα πρέπει να δούμε το θέμα του συντονισμού στην όλη τροφική αλυσίδα και την ιατρική τη διαδικασία και την ανθρώπινο παράγοντα. Και εδώ αυτό γίνεται κάπως περιφερειακά, ε, περιθωριακό σε σχέση με τη χρήση που γίνεται σε κτηνιατρικό επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ότι χρειάζεται να είναι η πρώτη προσέγγιση για να σώσουμε ό,τι μπορούμε. Και λέτε γιατί δεν προχωράει σε επενδύσει η βιομηχανία. Τι να σας πω, ε, δεν είμαι σε θέση να καταλάβω ορισμένα ηθικής φύσεως ε, σκέψη, ας πούμε γιατί κάνει η βιομηχανία ή όχι. Και αρκετές φορές κάπως μπερδευόμαστε και θα πρέπει να, μιλήσουμε γιατί θα πρέπει να πληρώνουμε δεκάδες χιλιάδες ευρώ για ένα φάρμακο ας πούμε για τον καρκίνο, για μια μορφή καρκίνου που δεν μας δίνει όμως και πολλά περιθώρια και καταλαβαίνετε ε, να σας πω όπως σύμφωνα με τις αρμοδιότητες μου δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα γι' αυτό αλλά ένα ίδρυμα με ρυθμιστικό χαρακτήρα τι μπορεί να κάνει να βρει τους κατάλληλους τρόπους για να προχωρήσει σε μια πολύ πιο γοργή εκτίμηση και να μειώσει οτιδήποτε έχει να κάνει με γραφειοκρατικό κόστος. Το τι μπορούμε να κάνουμε αυτό είναι και πρέπει να κάνουμε. Για να δούμε τώρα το περιθώριο κέρδους για τη μηχανία είναι εκτός αρμοδιοτήτων μας. Ναι. Νομίζω ότι πρόκειται για θέμα πολιτικό. Και εδώ με τους συναδέλφους χρειάζεται να το εξετάσουμε. Γιατί τι γίνεται. Παραμείνουν άλλοι τα προβλήματα δημόσιας υγείας πολύ σημαντικά. Και ίσως μέσω διαβουλεύσεων να δούμε, να συνονοηθούμε. Σας ευχαριστώ για το ανοιχτό πνεύμα που έχει το ανοιχτό κοινοβούλιο απέναντί μου και απέναντι στον οργανισμό. Και εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ο μόνο τρόπο να λύσουμε το πρόβλημα. Δηλαδή να υπάρχει μια πολύ συνεργασία μεταξύ ενό τεχνικού οργάνου που θα πρέπει να παρέχει όλα τα δεδομένα ε, τις γνώσεις για να μπορέσετε εσείς κατόπιν να τα μεταφράσετε στη νομοθεσία και στη συνέχεια εμείς θα θέσουμε αυτή τη νομοθεσία φυσικά σε πράξη και σε εφαρμογή. Σας ευχαριστώ. Bien. Πολύ ωραία. Ολοκληρώσαμε και το δεύτερο γύρο. Κερδίσαμε και χρόνο. Θα περάσουμε στο τρίτο γύρο. Τώρα έχουμε διαφορετικούς κανόνες. Έχουμε ένα λεπτό για τους βουλευτές και δύο λεπτά απάντησης για σας κύριε Διευθυντά. Δεν αλλάζει, αλλά δεν έχουμε δευτερολογία στην ερώτηση. Παρακαλώ. Κυρία Ριβάζη, ναι. Κύριε Υποψήφι εγώ θέλω να επανέλθω στην προστασία των ασθενών. Το προσεγγίσατε κάπως και θέλω να σας αναφέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα έχουμε κάποια εμβόλια που θέσαμε στην αγορά και μετά από ένα έτος είδαμε ότι υπάρχουν ε, παρενέργειες. Σε χάρη ότι είχαμε ναρκοληψία στα παιδιά όταν εμβολιάζονται με αυτό το Πανμέριξ ε, και η Σουηδία και η Φιλανδία ναι, έστειλαν ε, τον εμβολιασμό με τα προϊόντα αυτό γιατί είδαν ότι υπήρχε ουσιαστικά σύνδεση μεταξύ ναρκοληψίας και των εμβολίων αυτών και σήμερα η Τουρκία ανέστειλε τη χρήση των εμβολίων αυτών. Τι έκανε ο ΕΟΦ, δεν έχουμε ακόμη αρκετέ μελέτε, πρέπει να έχουμε και άλλε μελέτε και δεν ε, ε, να στέλνουμε τη χρήση αυτού του προϊόντο. Εγώ θέτω μια ερώτηση λοιπόν, αν υπάρχουν χώρε ε, που κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, γιατί, ε, μάλλον, ποια διαδικασία πρέπει να θέσουμε σε εφαρμογή για να πούμε ότι τελικά εφαρμόζουμε την αρχή τη πρόληψη για του ασθενού παρά ε, στα εργαστήρια. Έτσι λοιπόν, ε, ε, αντί, παραδείγματο χάρη αυτού του εμβολίου, εμβολίου έχουμε άλλο εμβόλιο όπως το έπρεπε και άλλα τα οποία επιτελούν την ίδια λειτουργία τελικά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ε, ξέρω, δεν μπορώ εγώ να πω ότι αν έδρασε σωστά ή όχι ο έφεγος, συμφωνώ μαζί σας. Ε, μπορούμε να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα από αυτά που συνέβησαν. Εγώ νομίζω ότι επιστρέφουμε στο πρόβλημα της φαρμακοεπαγρύπνησης ε, και στο πρόβλημα της ε, ε, κάπως γρήγορης θέσης εμπορία ορισμένων φαρμακών. Η επιταχυμένη διαδικασία, αν δεν υπάρχουν όπως έγινε στην περίπτωση της πανδημίας, ε, τότε ουσιαστικά εκεί υπήρχε επιβολή από τον ΠΟΗ, από οργανισμούς ανωτέρου παιδού. Είχαμε πολύ λίγο χρόνο για να αντιμετωπίσουμε μια, την έλευση μιας πανδημίας. Έτσι λοιπόν, ο ΕΟΦ έπρεπε να συντομεύσει ώστε να το περισσότερο της διαδικασίας αδειοδότησης. Αυτή είναι μια συζήτηση μεταξύ κινδύνου και ωφέλου. Ε, ε, δηλαδή πρέπει πάντοτε να βλέπουμε ποια είναι τα διδάγματα για το μέλλον. Εγώ τώρα ακόμη δεν έχω αναλάβει τα καθήκοντά μου στον ΕΟΦ ε, και δεν ξέρω για ποιο λόγο ΕΟΦ δεν σταμάτησε αυτή τη διαδικασία στην Ευρώπη. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει εποπτεία στην όλη διαδικασία και αυτό αφορά δύο πτυχές. Δηλαδή πρέπει να βλέπουμε και τα αριθμητικά στοιχεία αλλά θα πρέπει να αξιολογούμε και τις παρενέργειες γιατί σε ορισμένε περιπτώσεις ε, μπορεί να αποσύρουμε ένα φάρμακο το οποίο έχει όφελος. Βέβαια δεν ήταν αυτή η περίπτωση. Εγώ νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με την εφαρμογή στην οποία πρέπει να προβεί η αίμα, στην εφαρμογή όλων των διαδικασιών ε, ταχείας αξιολόγησης, ε, ε, των συνεγερμών της φαρμακοεπαγρύπνησης και των τρόπων αξιολόγησης του κινδύνου. Κύριε Διευθύντα, να θέσω κι εγώ μια ερώτηση γενικού χαρακτήρα για την ομάδα μου. Γράφετε στο πνεύμα όσων είπαν και συνάδελφοι, βιώσαμε διάφορες κρίσεις και όλοι αισθανθήκαμε και τη σημασία αλλά και την αναγκαιότητα μιας, ενός τέτοιου οργανισμού όπως ο δικός σας, ε, ως ένα όργανο που να μπορεί να είναι αρμόδιο να λάβει αποφάσεις ε, στην παιδοκρατών και ταυτόχρονα αναρωτιόμαστε για το βαθμό εμπιστοσύνης που μπορούμε να έχουμε. Δηλαδή, πώς ε, φαντάζεστε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε το επίπεδο εμπιστοσύνης στο δικό σας οργανισμό και πέρα από την δική μας εμπιστοσύνη και την εμπιστοσύνη των πολιτών. πιστεύω ότι το πρώτο επίπεδο της οικοδομής της εμπιστοσύνης ε, είναι της ε, διαχείρισης, είναι αυτό της διαχείρισης της, ε, των συγκρόμενων συμφερόντων των ανθρώπων που καλούνται τελικά να πάρουν τις τελικές αποφάσεις. Ο δεύτερος άξονας είναι αυτός της επικοινωνίας. Πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με την Κομισιόν και με το Κοινοβούλιο. Πρέπει να είναι στοχευμένη η επικοινωνία αυτή σε σχέση με το πώς ε, και γιατί λαμβάνονται οι αποφάσεις. Και πρόκειται για ένα επίπεδο επικοινωνίας που καθιστά τον ΕΟΦ την τεχνική πηγή της πληροφόρησης ε, πολύτιμων πληροφοριών. όπως ε, επίσης ε, και ως συναλλακτική πληροφοριών ε, έναντι παραπληροφόρησης που έρχεται από το δίκτυο και είναι όλο και πιο ενισχυτικό ότι πολλοί ασθενείς πληροφορούνται όλο και περισσότερο από τη διαδίκτυο και δεν υπάρχει συνεχής ροή πληροφοριών από την πλευρά των ευρωπαϊκών θεσμών που είναι αρμόδιοι για την υγεία και ο ΕΟΦ ε, βρίσκεται στη βάση αυτού. Πρέπει να επικοινωνεί άμεσα, αλλά θα πρέπει να παρέχει και σημαντικές πληροφορίε. Εγώ νομίζω ότι μόνο έτσι μπορούμε να πανικοδομήσουμε την εμπιστοσύνη και το τρίτο σκέλος αναφέρθηκε πολλές φορές, αλλά πρέπει να αναφερθούμε στο θέμα της διαφάνειας. Αν εμεί ανακοινώνουμε γιατί ε, λαμβάνονται οι μα ε, και ε, βάσει ποιες διαδικασίες. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στον πληθυσμό και θα ε, θεωρεί ότι ο EMA και οι υπόλοιποι οργανισμοί είναι ένα σημείο αναφοράς και ε, ένα σημείο πρόσβασης στη γνώση, συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τον τομέα της υγείας. Κύριε κύριος Περνιό. Ερώτηση. Το αλφακόλ ε, είναι ένα προϊόν ε, ε, το οποίο χρησιμοποιείται για νόσους του σηκωτιού και προήρθε από την έρευνα στα νοσοκομεία, στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία και η, μάλλον το... η εναλλακτική στο φάρμακο αυτό είναι στο να υπάρχει μεταμόσχευση ε, ύπατος. Ε, η... τέθηκε σε εμπορία ε, αυτό το φάρμακο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε άδεια, ε, μάλλον επέτρεψε αυτή την άδεια όμως ε, μια ε, άλλη εταιρεία ζήτησε να μην δοθεί η άδεια αυτή. Ε, πώς μπορούμε να αποκτήσουμε μεγαλύτερη διαφάνεια μεταξύ του δικού σας έργου, δηλαδή του ΕΟΦ, σε σχέση και με όσα κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μικρόφωνο παρακαλούμε. Μόνο εν μέρει γνωρίζω την περίπτωση αυτή. Ξέρω ότι πρόκειται για ένα φάρμακο που αποκαλείται ορφανό και το ανέκρινε η Κομισιόν, όμως η παθολογία αυτή αφορά περίπου 70 ασθενείς στην Ευρώπη. Ε, πρόκειται για ένα γενετικό πρόβλημα που προέρχεται από τη χολή. Και στην περίπτωση αυτή το πρόβλημα της πρόσβασης είναι σχετικό γιατί για παρηγορητικούς στόχους, για παρηγορητικούς σκοπούς ε, δίνεται η δυνατότητα σε ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε μια τέτοια θεραπεία. Νομίζω ότι τώρα μου δίνεται η ευκαιρία να επανέλθω στη σημασία της συνεργασίας και της αμοιβές εμπιστοσύνη. Είναι προφανές ότι είναι απαράδεκτο για τον εύστο μέλλον να λαμβάνει αποφάσεις ε, με τις οποίες δεν συμφωνεί η Κομισιόν, όχι επειδή θα φταίει η Κομισιόν, αλλά λόγω ελλείμματος επικοινωνίας ή εξοπιστίας. Και εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι το πρώτο σημείο επί το οποίο θα πρέπει να εργαστώ, έτσι ώστε να υπάρχει απόλυτο ε, συντονισμό ε, θεωρήσεων και προθέσεων και να υπάρχει απόλυτη αξιοπιστία του έργου τη CMA, η οποία έχει όλη την εμπειρογνωμοσύνη για να μπορεί να διαλογίσει τι αποφάσει που λαμβάνει. Ευχαριστώ, κυρία Μπέρεντ. Uh, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κύριε Ράζη, συμφωνείτε μαζί μου στο ότι πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των δύο διαδικασιών. Αφενός δηλαδή όπου υπάρχει ευθύνη τη ΕΟΦ και από την άλλη των κρατών μελών και να μην τα μπλέκουμε. Και μετά ένα ερώτημα για την ασφάλεια των ασθενών. Τι θέλουμε να κάνουμε στις περιπτώσεις όπου αφενός έχουμε την ε, τεράστια ζήτηση φαρμάκων από τους ασθενείς και από την άλλη δεν είμαστε απολύτως σίγουροι πως είναι ασφαλές ένα φάρμακα. Μπορώ να σας απαντήσω κι εγώ. Δεν υπάρχουν, ήδη, δεν υπάρχουν 100% ασφαλή φάρμακα και πρέπει να μην έχουμε αυτή την ψευδέστηση. Δεν πρέπει να παριστάνουμε ποτέ κάτι τέτοιο. Τα φάρμακα πάντα έχουν κάποιον κίνδυνο και ο κίνδυνος αυτός πρέπει να είναι μικρότερος από το καλό που κάνουν. Και όταν το καταφέρνουμε αυτό, τότε κάνουμε καλό. Συμφωνείτε με αυτό, έστω και ελαφρώς, κύριε Ράζη. Σε ό,τι αφορά τώρα τις εθνικές διαδικασίες, το δίχως άλλο δεν μπορούμε να μην σεβαστούμε ορισμένους ε, εθνικούς κανόνες που σχετίζονται με συνήθειες ζωής, ε, με την παράδοση, με την οικονομική και κοινωνική κατάσταση. Σας υποστηρίζω σε αυτό, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι εκεί όπου υπάρχει δυνατότητα εναρμόνισης και όπου η εναρμόνιση θα επιφέρει όφελος για τους πολίτες, πρέπει να την επιδιώξουμε την εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τώρα το πρόβλημα της ασφάλειας των φαρμάκων, αν μπορώ να το περιγράψω έτσι, θα σας πω μια εντύπωση που είχα πριν 7-8 ε, χρόνια, όταν για πρώτη φορά μπήκα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Τελικού Οργανισμού. Αισθάνθηκα σαν ένα άτομο που είχε δύο πιστολιά στο κρόταφο, έναν από τους ασθενείς που ήθελαν το φάρμακο αυτό αμέσως και το άλλο από τους ίδιους ασθενείς που έλεγαν ότι αν βάλω το φάρμακο αυτό στην αγορά, το θέσω στην αγορά, είμαι φιλός της βιομηχανίας. Ε, είναι σχιζοφρενική η θέση αυτή και πράγματι είναι μια θέση ε, η οποία ε, ουσιαστικά εξηγένεται μόνο ε, αν ακολουθήσουμε αυστηρά την επιστήμη. Πρέπει δηλαδή να βασίζουμε τη γνώση μας σε όσο το δυνατόν περισσότερες αποδείξεις. Πρέπει να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερες τεχνικές μελέτες, τις καλύτερες τεχνολογίες που μας επιτρέπει τώρα η επιστήμη σε ό,τι αφορά τους βιοδείκτες ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν κλινικής απάντησης που ε, να προβλέπει τις παρενέργειες του φαρμάκου. Το φάρμακο ονομαζόταν δηλητήριο από τους Έλληνες. Έτσι λοιπόν, ας ε, μην ξεχνάμε ε, ότι ήταν η μετάφραση στα Ιταλικά του όρου φαρμάκου ήταν η λέξη δηλητήριο. Έτσι λοιπόν, κάθε φάρμακο μπορεί να έχει και μια σκοτεινή πλευρά. Εμείς αξιολογούμε το θέμα του κινδύνου ε, ε, και φυσικά δεν μπορούμε να υπονομεύουμε τον κίνδυνο, να μειώνουμε τον κίνδυνο. Κύριε Γκαρντίν, ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ, Πρόεδρε, ευχαριστώ, κύριε Ράζη. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που εσείς θίξατε σε μια άλλη απάντηση για το διαδίκτυο. Έχετε δίκιο, εμεί βλέπουμε τα δεδομένα, Μα λένε ότι οι πολίτες ε, στρέφονται λένε και περισσότερο στο ίντερνετ ε, και ε, για ενημέρωση αλλά και για αγορά φαρμάκων και είναι η κύρια πύλη εισόδου των ψευδεπίγραφων φαρμάκων και μάλιστα μπορούν οι ασθενείς έτσι να έχουν πρόσβαση και σε φάρμακα χωρίς συνταγή. Είναι σοβαρό θέμα αυτό λοιπόν για την υγεία. Θα ήθελα εσεί να μου πείτε τι σκέφτεστε σχετικά και ποια στρατηγική θα μπορούσε να αναχαιτήσει το φαινόμενο αυτό το οποίο αν το εγκαταλείψουμε όσο έχει από ό,τι φαίνεται θα αυξηθεί γιατί με τη διάδοση τεχνολογιών και με τις νέες γενιές που χρησιμοποιούν όλο και περισσότερο το διαδίκτυο εμείς ε, θα δούμε ότι αυτό το φαινόμενο θα έχει θεαματική αύξηση τα επόμενα έτη. Ναι, ευχαριστώ. Πράγματι το διαδίκτυο είναι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του πολιτισμού και ένα από τα μεγάλα προβλήματα. Η ιατρική ενημέρωση, οι ιατρικές πληροφορίες έρχονται όλο ένα και περισσότερο μέσω του διαδικτύου και από πηγές που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Το αδύναμο σημείο στην Ευρώπη το πρόβλημα της πλαστογράφησης των ε, φαρμάκων είναι σχετικά χαμηλό των πλαστών φαρμάκων. Ε, στην Ιταλία είναι 0,01 γιατί έχουμε και ένα πολύ αποτελεσματικό δίκτυο διανομής ε, και δεν υπάρχουν φάρμακα online. Είναι παράνομα δηλαδή, αλλά πραγματικά από εκεί μπορούν να μπουν τα ψευδοεπίγραφα φάρμακα. Τα φάρμακα αυτά απειλούν την υγεία, αποτελούν κίνδυνο για την υγεία Τώρα, τι έχει γίνει. Έχουμε ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο λέγεται Impact. Συμμετέχουν πολλά κράτη και ο ΕΟΦ, αν δεν το κάνει νομίζω ότι θα συμμετέχει αν εξαρτηθεί αυτό από μένα. Το μεγάλο πρόβλημα ε, σίγουρα το κοινοβούλιο έχει, ε, είναι ένα από τα καταλαβήματα για να επιληθεί το πρόβλημα είναι να κάνουμε εδώ μια αναβαθμίση του επίπεδου ε, ολοκλήρωσης ε, δηλαδή πρέπει εδώ να συμμετέχει και η αστυνομία πρέπει να έχουμε στρατηγικές πληροφορίες και πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να ελέγχουμε το διαδίκτυο στην Ευρώπη. Κατασχέθηκαν πέρσι 25 τόνοι δραστικών ουσιών ε, πλαστών που προέρχονταν από την Ασία. Χάρη σε αυτό το project, το Impact, ε, το οποίο ε, ελαφρώς χρηματοδοτήθηκε από κάποιες εθνικούς οργανισμούς και δεν υποστηριχθήκε ιδιαίτερα. Χρειάζεται μεγαλύτερο συντονισμός και ρυθμιστικός οργανισμός φυσικά αναλαμβάνει αυτή τη δράση. Peter pour la dernière question. για την τελευταία ερώτηση. Ja, vielen Dank nochmal. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε υποψήφιο διευθυντά, έχω μια ερώτηση για τους εκπροσώπους των ασθενών το Κοινοβούλιο. Πάντα έλεγε να εκπροσωπούνται και εκπρόσωποι των ασθενών στα φόρουμ της, του ΕΟΦ, αλλά δεν έχουμε ακόμα με επαρκή χρηματοδότηση. Βεβαίω είναι επικριτικό όταν μια συγκεκριμένη εταιρεία χρηματοδοτεί μια οργάνωση, τότε προφανώς εκπροσωπεί τη βιομηχανία περισσότερο, αλλά την άλλη δεν υπάρχουν άλλες δυνατότητες χρηματοδότησης. Θα μπορούσατε να μας υποβάλλετε κάποιες ιδέες, προτάσεις για το πώς θα έχουμε ανεξάρτητη χρηματοδότηση οργανώσεων ασθενών και όχι μόνο τους συνήθεις κάθε φορά αλλά και για αυτούς οι οποίοι κάθονται στα διάφορα φόρουμ. Κύριε Διευθυντά, θα μπορούσατε να απαντήσετε την ερώτηση αυτή και μετά ολοκληρώνουμε. Παρακαλώ, 5 με 6 λεπτά. Ναι. Σας ευχαριστώ. για τις ένωσεις των ασθενών και το πώς συμμετέχουν και για τη χρηματοδότηση βέβαια. Είναι ιδιαίτερο ευρύ το πρόβλημα, όπως ακριβώς για τη χρηματοδότηση της έρευνας και για την ανεξαρτησία διαφορών ερευνών. Θα μπορούσε να αποτελέσει μια λύση το να έχουμε ταμεία, την σύσταση ταμείων μια ένωση ασθενών ακριβώς να χρηματοδοτείται από ένα θωρακευτικό εργαστήριο και μετά από τη στιγμή που ενδιαφέρεται ακριβώς από τις ενδείξεις αυτές τις ασθένειες και τα συμπτώματά τους κλπ. Να συσταθεί ένα ταμείο κατά ορισμένου όρου και να μην ξέρει κανεί τελικά πού θα κατευθυνθεί αυτή η χρηματοδότηση. Και αυτό για τα ποσά που τα κονδύλια που μας έρχονται από την ίδια τη βιομηχανία. Εντάξει, ένα κάποιο ποσοστό τόσο της εκατό ή τόσο της χιλής ας πούμε κάπου για τη χρηματοδότηση αυτή και να χρηματοδοτεί τις σχετικές δραστηριότητες ώστε να μην ε, συνδυάζεται με βιομηχανικό ενδιαφέρον ε, του εργαστήριο αυτό. Πολλές φορές οι ασθενείς ε, δεν γνωρίζουν αλλά προκαλούν, δημιουργούν, ελκύουν το ενδιαφέρον της βιομηχανίας. Στην που δεν θα είναι κρατικά κονδύλια, μόνο ένα γενικό ταμείο που θα μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση θα μπορούσε τώρα άμεσα να αποτελέσει μία λύση. Η γενικής φύσεως συμπεράσματα τώρα. Αρκετά είπαμε για, για πάσης φύσεως προβλήματα Ελπίζω να είμαι και ο σωστός άνθρωπος ε, για την εντολή αυτή, για τη θέση αυτή. Στον ΕΟΦ έχουμε ε, μια ευρή ομάδα, ακριβώ χρειάζεται και καλύτερο συντονισμός. Χρειάζεται να αλλάξουμε και στο μέλλον μερικά πράγματα. Χρειάζεται να αλλάξει η όλη εικόνα της δημόσιας υγείας και της παρασκευής φαρμάκων. Είναι κάτι που συνεχώς μεταβάλλεται. Πριν από δύο χρόνια αυτό που ίσχυε σήμερα δεν νομίζω να ισχύει. Δεν θα μπορούσα να το επαναλάβω. Τα ευρωπαϊκά ε, συστήματα υγείας ε, ε, νομίζω ότι εντάξει κάπως εξασφαλίζουν την υγεία στους πολίτες, αλλά υπάρχει ακόμα περιθώριο για να βάλουμε τα πράγματα σε μια αυθολογική βάση, για καλύτερες επενδύσεις και να έχουμε ακόμα περισσότερη υγεία για τους Ευρωπαίους πολίτες. Ασχοληθήκαμε με αρκετά θέματα, δεν ξέρω, δεν μου έρχεται τίποτα άλλο συγκεκριμένο στο μυαλό για να σας προτείνω, αλλά οπωσδήποτε Εάν θέλετε μια κάποια περαιτέρω διευκρίνηση θα μπορούσα να σας απαντήσω και ελπίζω να μπορέσω να συνεχίσω την επαφή μαζί σας και να βοηθηθούμε εδώ και στην, ε, στην αίθουσα αυτή, στην Επιτροπή σας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή που μου αφιερώσατε. Κύριε Διευθυντά, εξ ονόματος των συναδέλφων, ε, σας ε, ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας ε, σε όλους. Με πολλά θέματα ασχοληθήκατε και μας διαφορετικής φύσης απόγευμα και απαντήσατε σαφώς με διαφάνεια, σαφήνεια και απαντήσατε έτσι λοιπόν. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα γιατί ανταποκριθήκατε σε αυτό το έργο. Ε, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι μια εύκολη δουλειά και απλή για σας. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Πέρα στις συνεδρίες. La réunion des coordinateurs aura lieu à 10. η ώρα συντονιστές.